Συμβουλίου ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτή και σε ό,τι αφορά την ε, ανακοίνωση των προτάσεων διάσκεψης του Προέδρου για τους ορισμούς στις κοινοβουλευτικές επιτροπές πρέπει να σας πληροφορήσω ότι θα σας διαβιβαστούν όλα αυτά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο ίδιος κατάλογος θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά της σημερινή συνεδρίασης και επίσης πρέπει να σας πω ότι η προθεσμία κατάθεσης ε, ε, τυχών τροπολογιών ολοκληρώνεται απόψε στις 7. Η δε ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 9 το πρωί, στην αρχή της συνεδρίασης. Σας εύχομαι καλό σας βράδυ και ε, τη διακοπή της συνεδρίασης.